Καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να μην παγιδεύτηκε κανείς από τη φωτιά που ξέσπασε. Γιατί εγώ κλείστηκα κάπου, ε, έπεσε μια πόρτα μπροστά μου και έπρεπε να φύγω από άλλο σημείο. Μπορεί να έρθουν άλλη ώρα οι συνάδελφοι. Αρχίζει η απογευματινή συζήτηση με τις συμβαστικές τροπολογίες του κυρίου Ροσφόρ για την έκθεση προφανώς του κυρίου Ροσφόρ, πρόγραμμα καταναλωτές για την περίοδο 14-20. Παρευρίσκονται οι σκιώδη Σάιμον Μπούσουτλ και η Μαρία Ιριγκόγεν Πέρες. Η Χάιντε Ρούλε απουσιάζει ακόμα και οι υπόλοιποι δεν ξέρω επίσης θα καταφτάσουν φαντάζομαι. Και εγώ είμαι εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, και χαίρομαι που βλέπω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μάινερ ήθελε να είναι παρούσα, αλλά το πρωί περίμενε και κάθισε μια μισή ώρα για το ADR και προφανώς έχει και άλλες δουλειές η γυναίκα, δεν θα καθόταν εδώ όλη μέρα. Ο κύριος Ζωσφόρ έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει συμβαστικές τροπολογίες. Ναι, θα ήθελα να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Την τελευταία φορά σας είχα πει ποια ήταν η απόψή μου για μεμονωμένες τροπολογίες. Βρισκόμαστε τώρα στην τελική όμως φάση γιατί αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τους ε, συναδέλφους μου οι οποίοι πραγματικά με υποστήριξαν πολύ στην όλη μου προσπάθεια. Είχαμε πραγματικά μια, ένα εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας. Καταφέραμε επίσης να σωματώσουμε και κάποιες νέες ιδέες και καταλήξαμε τελικά σε 11 συμβαστικές τροπολογίες. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε πάρα πολλά σημεία. Επί τη ουσία δεν ήταν δύσκολη η δουλειά μα άλλωστε. Συναντήσαμε κάποιε δυσκολίε γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια πολύ τεχνικά σημεία. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να έχει απόλυτη αυστηρότητα και συνεκτικότητα. Το ΕΛΚΑ, οι Σοσιαλδημοκράτες και το ΑΛΔΕ συμφώνησαν για συγκεκριμένε τροπολογίες και οι πράσινοι όμως κατάφεραν να μας υποστηρίξουν, οι ίδιοι όμως δεν είχαν υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω εντάχει τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Δεν θα σας παρουσιάσω τις συμβαστικές τροπολογίες ξεχωριστά, αλλά τις βασικές ιδέες επί των οποίων καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Πρώτον, μιλήσαμε εκτενέστατα για έναν σαφέστατο στόχο, να υποστηρίξουμε τις δράσεις εκείνες που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον καταναλωτή να διαδραματίσει καλύτερα το ρόλο του στην εγχώρια αγορά. Υπήρχε το θέμα της συγκρισιμότητας των δεδομένων για να έχουμε μία διαφάνεια στην αγορά και επιμείναμε στο ότι δεν τίθεται μόνο το ζήτημα των τιμών αλλά και της ποιότητας για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πηγαίνουν προς τον καταναλωτή. Ένας προετοιμασμένος καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει και την τιμή αλλά και την ποιότητα του προϊόντος. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να υπάρχει η απαραίτητη αυτή σήμανση και να αναφέρεται σήμανση αυτή και το σελίδε εκείνες οι οποίες συγκρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να ισχύουν ε, μέθοδοι εναρμονισμένες για τη σύγκριση αγαθών και υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να ισχύει ο κανόνας αυτός προκειμένου να μπορούμε ανοιχτά να συγκρίνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στην εσωτερική αγορά και κατά αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούμε καλύτερα και ποια είναι η δυναμικότητα, η δυναμική της εσωτερικής αυτής της αγοράς. Δεύτερο σημείο που το οποίο συμφωνήσαμε είναι η κατάρτιση, η πληροφόρηση, η ενημέρωση των καταναλωτών. Εκπαίδευση καλύτερα των καταναλωτών. Όντως υπάρχουν ευπαθή άτομα, ευάλωτα άτομα, τα οποία προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε μέσω, των, μέσω της καρτάρτισης των ε, καταναλωτών, της διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών. Ξέρετε ότι ε, είμαστε καταναλωτές στη σημερινή κοινωνία από την ημέρα της γεννησής μας ε, μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής μας. Και μια άλλη ιδέα που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν το να συμμετέχουν και επιχειρήσει στη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών. Αυτό μα προκαλεί μερικέ φορέ εντύπωση, αλλά πραγματικά αν καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε μια επιχείρηση, τότε τα πράγματα λειτουργούν πάρα πολύ θετικά. Υπάρχει μια θετική μόχλευση. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιχείρηση να μπορεί να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή, με απόλυτη διαφάνεια. Όσον αφορά τώρα τους ευπαθείς, ευάλωτους καταναλωτές, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και τροπολογίε που είχαν ω στόχο ακριβώ να βοηθήσουν αυτού του καταναλωτέ. Ένα άλλο σημείο που το οποίο δεν είχαμε απόλυτα συμφωνήσει ήταν για τον ε, ρόλο που θα έπρεπε να λάβουν οι καταναλωτέ και το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την υποστήριξη των δράσεων υπέρ των καταναλωτών. Σα υπενθυμίζω και νομίζω ότι συμφωνούμε από αυτού ότι ε, η άμεση χρηματοδότηση για τις ε, οργανώσεις θα πρέπει να γίνει για τις οργανώσεις εκείνες που είναι διασυνοριακές, ευρωπαϊκό δηλαδή επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τις ε, εθνικές ενώσεις καταναλωτών που βρίσκονται σε κάθε κράτος μέλος. Η βοήθεια όμως αυτή δεν θα πρέπει να λάβει τη μορφή άμεσης χρηματοδότησης. Είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διοργανική τους ικανότητα να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους και είπαμε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη όσον αφορά την έρευνα σχετικά με την κατανάλωση που θα έχει ως στόχο να βοηθά τους καταναλωτές και να λειτουργεί προς το συμφέρον των καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση του προγράμματος και τη συνέχεια θα, θα πρέπει να δοθεί. Πάλι εδώ πέρα εντοπίσαμε πολλά ευαίσθητα ζητήματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από τις κατεξοδότηση πράξης όσον αφορά τετήσια προγράμματα, καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποιους συμβασμούς όσον αφορά τους δείκτες που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε καλύτερα τα προγράμματα αυτά. Και υπήρχε ένα άλλο σημείο το οποίο οδήγησε σε έντονες συζητήσεις, δηλαδή το ζήτημα της κατανομής των πόρων που θα πρέπει να δοθούν σε κάθε στόχο. Έγινε λοιπόν μια έντονη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατανομή της χρηματοδότησης στο παράρτημα 2, το οποίο έχουμε στο νομοθετικό μας κείμενο. Ουσιαστικά είναι ένα ενδεικτικό κείμενο. Είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα περιθώριο ευελιξίας αναφέρομαι στις τροπολογίες 73 και 74, ένα περιθώριο της τάξης του 20 περίπου της 100 και μία ακόμα συμβαστική πρόταση που έγινε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δείχνουμε ουσιαστικά ότι θέλουμε να έχει ένα περιθώριο ευελιξία στα πλαίσια μια προφορική τροπολογία, βάση αρχική τροπολογία, προσθέτουμε το ότι θα πρέπει να υφίσταται η αναγκαία ευελιξία, την οποία θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε, εφόσον χρειαστεί, να έχει τη δυνατότητα να απομακρυνθεί από το αρχικό κείμενο που προβλέπει μια συγκεκριμένη ευελιξία, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η τροποποίηση αυτή των γραμμών του προπολογισμού που θα μπορέσει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τυχαίνει μια δικαιολόγηση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό μέσω των πράξεων κατεξοδότηση. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να συνοψίσω τις συμβαστικές αυτές ε, τροπολογίες, οι οποίες πιστεύω ότι μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Ευχαριστώ. Well, thank you. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μόλις κοίταζα τις νομοδοτήσεις και των άλλων επιτροπών και θα ήθελα στη συνέχεια να σχολιάσω μερικά σημεία τους. Για να δούμε ποιες μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι και της Νομικής Επιτροπής και του Προϋπολογισμού. Στο μεταξύ να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση μέχρι τις 3.30. Βλέπω και τη Χάιντι Ρούλα, ο Σάιμον Μπουσουτήλ και μετά η κυρία Ριγκόγεν και στη συνέχεια η Χάιντι Ρούλα. Uh, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ροσφόρ για την παρουσίαση που έκανε, για όλη την εργασία του για το ζήτημα αυτό και ιδίω για το πνεύμα συνεργασία το οποίο κατέδειξε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο στην παρέμβασή μου. Θα έλεγα ότι το ΕΛΚ είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις συμβαστικές τροπολογίες του συμβασμού στου οποίου έχουμε καταλήξει μέσω διαπραγματεύση, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί έδειξε ιδιαίτερη διαλλακτικότητα όσον αφορά κάποια εκκρεμή ζητήματα για μας τουλάχιστον για το ΕΛΚ, όσον αφορά την κατανομή των στόχων 1 και 2, τη χρηματοδότηση για τους στόχους αυτούς. Δεν συμφωνώ με την ανακατανομή των ενδεικτικών ποσών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. παρόλα αυτά μπορώ να υποστηρίξω την άποψή του, αρκεί να υπάρχει μια αυξημένη ευελιξία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στην ουσία δεν θα περιορίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα ενδεικτικά ποσά. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να τονίσω έχει να κάνει, την, έχει να κάνει με τροπολογία 122 την οποία υπεβάλαμε. Πρόκειται για μια τροπολογία η οποία ζητά να δοθεί απαραίτητη σημασία και προσοχή στους ανήλικους, δηλαδή να μην έχουμε παραπλανητικές επιθετικές διαφημίσεις οι οποίες να απευθύνονται στους ανήλικους είτε στις τηλεοράσεις είτε online στο διαδίκτυο. Αναφίβολα ευπαθής ομάδα καταναλωτών είναι και τα παιδιά και οι ανήλικοι Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις ομάδες αυτές και τα καταναλωτικά τους δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν και άλλες πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία την 122, την οποία δεν επιθυμώ να αποσύρω. Του των λεχθέντων πιστεύω ότι μετά την αυριανή ψηφοφορία θα έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο συγητή στι διαπραγματεύσει που θα κάνει με το Συμβούλιο για το πολύ αυτό σημαντικό ζήτημα. Κατά την άποψή μου υπήρξε ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες και επομένω πιστεύω ότι ο εισηγητή θα έχει μια πολύ ισχυρή πολιτική θέση όταν θα μα εκπροσωπήσει στι διαπραγματεύσει που θα κάνει με το Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ριγκόγεν Πέρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μπούσουτιλ. Ευχαριστώ τον κύριο Βοσφόρ ε, ε, για ε, την προθυμία του και το οικοδομητικό πνεύμα της συνεργασίας. Κατανοώ την ευαισθησία του για τους ευάλωτους καταναλωτές και για άλλα θέματα που για τη δική μου πολιτική ομάδα είναι σημαντικά. Ε, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικές τροπολογίες και είναι πρωταρχικής σημασίας. Καταρχάς, άρση των εμποδίων άμεσων και έμεσων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών για να κάνουν διασυνοριακές αγορές. Επίσης, υποστήριξη των ε, οργανώσεων καταναλωτών με μηχανισμούς χρηματοδότησης για να ε, μπορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δρούν οι οργανώσεις καταναλωτών, το λέει και αυτό ο κύριος Ροσφόρ, και να ενισχυθούν ε, και σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό, σε εθνικό και ευρωπαϊκό, ε, με στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια που είναι απαραίτητη για να δοθεί μια όθηση και δυναμική στην εσωτερική αγορά. Βέλτιστες πρακτικές ενημέρωση καταναλωτών και έρευνα αγοράς είναι πολύ σημαντικά για την κατανάλωση ανάπτυξη και ενίσχυση επίσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της δυνατότητας ε, να κάνουν εύκολα, γρήγορα, φθηνά παράπονα και καταγγελίες. Στη συνέχεια, ανάγκη εποπτείας και αξιολόγησης των μέτρων του προγράμματος για να γνωρίζουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων και να αποφύγουμε τις τρευλώσεις ε, στη λειτουργία της αγοράς. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου που στις συμβαστικές τροπολογίες δεν έχετε συμπεριλάβει το ζήτημα της συμμετοχής ε, καταναλωτικών οργανώσεων στην πρακτική οργάνωση των συστημάτων επίλυσης διαφορών. Όπως επίσης δεν προβλέπεται και χρηματοδοτική ε, βοήθεια. Και ζητώ συγγνώμη γιατί συζητιέται έκθεσή μου σε άλλη επιτροπή στην Περιφερειακή και πρέπει να φύγω για να πάω εκεί. Ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ. Okay. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, έτσι κι αλλιώς ε, ξέρω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας είναι υπερδραστήρια και εργάζονται κι άλλο. Ευχαριστώ. Κύριε Ρούλε, ε, μπορεί να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ε, γράψαμε στον ε, εισηγητή. Είναι πολύ καλή η έκθεσή σας. Την υποστηρίζουμε. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. ευχαριστώ. Yeah. Uh, well, as the last shadow rapporteur before we get on. τελευταίο μπορώ να πω το ίδιο. ως τελευταίο σκιώδη συζητητή, ότι θα υποστηρίξουμε αυτές τις προτάσει συμβιβασμού. Η κυρία Κοξεμπίπ θα ήθελα να πάρει το λόγο. Υπάρχουν, υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να μιλήσει, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ για την θαυμάσια δουλειά που έχει γίνει και θα ήθελα να υποστηρίξω τα όσα είπε ο Σάιμον. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 122 θα ήθελα να διευκρινίσω ένα-δύο πράγματα γιατί πιστεύω ότι μολονότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την ελευθερία του ίντερνετ για την ελευθερία έκφρασης στο ίντερνετ και να διευκολύνουμε ε, όλες τις καινοτόμους πτυχές ε, του ίντερνετ είναι πάρα πολύ σημαντικό παράλληλα με τους διάφορους φορείς ε, και την επιχειρηματική κοινότητα να έχουμε μία υπεύθυνη στάση σε ό,τι αφορά την εμπορία μέσω του ίντερνετ. Όλοι μας είμαστε γονείς και πραγματικά έχουμε ένα προβληματισμό ότι το ίντερνετ και μερικά από τα multimedia, από τα πολυμέσα στα οποία έχουμε πρόσβαση όλο και περισσότερο θα μπορούσαν να, έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε θέματα όπως η παχυσαρκία, το σεξ, ε, το χρήση, κατάκτηση νοπνεύματος κτλ θα, μήπως ο Ρομπέρ θα ήθελε λίγο να με ακούσει. Θα είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγουμε τη ρύθμιση του θέματος του διαδικτύου. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει υπεύθυνη διαφήμιση και αυτό ακριβώ ζητάμε εδώ. Στην ουσία δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεται το πρόβλημα στο να γράψουμε. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση των ανηλίκων και εξασφαλίζει την υπεύθυνη ε, διαφήμιση είναι η πιο φιλελεύθερη διατύπωση που θα μπορούσα να φανταστώ και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ της 120 δίνω γιατί δεν έχει καλυφθεί από τροπολογία συμβιβασμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος, και δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο και μετά θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμεί θα θέλαμε με τη σειρά μα να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή για την εξαίρετη αυτή έκθεση και για τι ε, τροπολογίε συμβιβασμού. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα σχόλια που θα θέλαμε να κάνουμε και για τα δύο. Ξέρετε την άποψη της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του ετήσιου προγράμματος. Κατά την άποψή μας αυτό δεν είναι το πλέον κατάλληλο μέσο. Παρόλη την ελαστικότητα, τη μείωση των δαπανών αναστόχο, πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην στη νομική πράξη, αλλά θα πρέπει να παραμείνει στις ε, δημοσιονομικές καταστάσεις όπως προτείναμε. Ε, σε ό,τι αφορά τις ιστοσελίδες συμφωνούμε απόλυτα για την κομβική σημασία που έχουν. Αυτό είναι κάτι που τονίζεται ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τον καταναλωτή αλλά έχουμε σοβαρότατο προβληματισμό σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ενός συστήματος πιστοποίησης που αφορά την εφαρμοσιμότητα του ελέγχου και της πιστοποίησης όλων των συγκρίσιμων ιστοσελίδων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό έχουμε, όπως σας είπα, έντονο προβληματισμό. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για μας. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να ε, υπάρχει κατάρτιση των επιχειρήσεων, αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα καταναλωτών που απευθύνεται σε καταναλωτές με πολύ μικρό ε, ε, προϋπολογισμό. Ένα μέρος του προϋπολογισμού θα δοθεί για την εκπαίδευση των επιχειρήσεων. Υπάρχουν βεβαίως και προγράμματα που έχουν ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Δέκα φορέ μεγαλύτερο από τον προπολογισμό των καταναλωτών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν τα λιγοστά κονδύλια που έχουμε εδώ θα πρέπει να δοθούν στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων, μόνο ότι συμφωνούμε με το γενικότερο στόχο. <clears throat> Αυτό είναι ένα θέμα ελάσσονο σημασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διατύπωση για την οργάνωση των καταναλωτών και για την άμεση χρηματοδοτική υποστήριξη, θα πρέπει να πω ότι το σημείο 112 σχετικά με την διαφήμιση στη τηλεόραση. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μιλάμε για ένα, δημοσιο... για ένα ε, οικονομικό πλαίσιο. Ποιος είναι ο αποδέκτης, σε τι πλαίσιο κινούμεθα. Όταν ε, παραθέτουμε την δράση αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της δράσης. Να προσέξουμε τι. Δεν είναι δράση αυτό. Ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα εκτιμώντας ε, θα μπορούσε να, θεωρη, να, θεωρηθεί ότι ανήκει σε μια γενική δράση, αλλά δίχως άλλο δεν είναι μια δράση που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτό το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο αποδέκτη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ενταχθεί αυτό στο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Δεν θέλω να παρατείνω, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Υπάρχουν και μερικά μικροσχόλια για τη διατύπωση. Πιστεύω όμως ότι αυτά είναι θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της γενικής συζήτησης με το Συμβούλιο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. πριν από την ψηφοφορία. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για τις γνωμοδοτήσεις ε, που λάβαμε και ποιες είναι οι τροπολογίες που θα σας έβρισκαν σύμφωνο. Ε, ευχαριστώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα λέγω ότι συμφωνούμε κατ' ουσία ε, με όλα. Νομίζω ότι η πρώτη σας παρατήρηση ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Πρόκειται για μία προφορική τροπολογία που αφορά τη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων. Ό,τι αφορά την τροπολογία 122 δεν θα πρέπει να κάνουμε λάθος. Συμφωνούμε απόλυτα σε ό,τι αφορά θέματα ουσίας αρκετά χρόνια χρημάτισα μέλος της Επιτροπής Εδεοντολογίας της Διαφήμισης. Ξέρετε ότι διέπεται ο τομέας αυτός από το καθεστώς αυτορύθμισης. Δηλαδή πολλοί επαγγελματίες ε, επιλέγουν το καθεστώς αυτορύθμισης. Συμφωνούμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την ουσία έχουμε κάποιο προβληματισμό σε ό,τι αφορά δύο σημεία. Το πρώτο σημείο, στο οποίο το, ε, το οποίο έθιξε ο πρόσωπο τη Επιτροπή, δηλαδή πρόκειται για ένα κείμενο που παραθέτει, που απαριθμεί τα προγράμματα. Και δεν ε, είναι σαφέ πώ θα μπορούσε αυτό να αντιστοιχίσει σε ένα πρόγραμμα. Και το δεύτερο, το δεύτερο σημείο που μας προβληματίζει είναι το θέμα τη εγγύηση των πρακτικών αυτών. Πώς θα μπορούσε η Επιτροπή να εγγυηθεί. Η λέξη εγγύηση είναι αρκετά έντονη, ενδεχομένω, είναι πρόβλημα γλωσσικό, ίσως η μετάφραση δεν έχει γίνει σωστά στα γαλλικά σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Κοιτάξτε, στα γαλλικά χρησιμοποιείται η λέξη guarantee, ε, που εγγυάται πρακτικές. Εγγυώμαι σημαίνει ότι βάζουμε μια σφραγίδα, δίνουμε μια εγγύηση ότι η διαφήμιση κτλ. Ενδεχομένως εκεί εγινε η δυσκολία. Αυτό που θα σας πρότεινα εγώ είναι να δούμε ενδεχομένως με την Επιτροπή εάν θα μπορούσε να γίνει κάποια προσαρμογή σε ό,τι αφορά τη διατύπωση, σε ό,τι αφορά το θέμα ουσία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Κατά κάποιον τρόπο όμω, αν θέλουμε να εγγυηθούμε πρακτικέ υπεύθυνη διαφήμιση, θα πρέπει να γίνει ένα ρυθμιστικό κείμενο, ένα νομοθετικό κείμενο που να διέπει τον τομέα τη διαφήμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ή θα δούμε ε, τι όρο θα επιλέγαμε, να μην είναι ένας τόσο ε, ισχυρός όρος ή θα δούμε αν θα, ή θα, μπορούσαμε να το ελέγξουμε ε, σε ένα εκτιμώντας, αλλά επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά θέματα ουσία συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχουν προτείνει οι άλλες επιτροπές, ε, κατά την προπαρασκευή του καταλόγου ψηφοφορίας όλα αυτά αναφέρονται σαφώς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα μείζωνος σημασίας. Αύριο θα ψηφίσουμε το σύνολο ε, και θα ήθελα απλώς να σας πω ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουμε γνωμοδοτήσεις που είναι πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει μετά το αποτέλεσμα του ε, ψηφοφορίας να κάνουμε μία επαλήθευση. Και εγώ θα πρότεινα να δούμε σε τι βαθμό θα, μπορού, θα ήταν ενδεχομένω σκόπιμο να προτείνουμε στους διονυστές της Επιτροπής ε, να ξεκινήσουν προπαρασκευαστικές συζητήσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος. Βεβαίως, μην ξεχνώντας ότι σε μία πρώτη φάση δεν θα γίνει μία αναφορά στο ποσό των συγκεκριμένων δράσεων. Θα πρότεινα να το δούμε αυτό μετά την αυριανή ψηφοφορία. Okay. Well, thank you. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν ότι ψηφίζουμε αύριο το πρωί από τις 9.30 και μετά και στη συνέχεια εναπόκειται στον εισηγητή να δει ποιες θα είναι, ποια θα τα επόμενα βήματα της στρατηγικής, όπου θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον προπολογισμό. Όπως είπατε, υπάρχει και ένας συγκεκριμένος χρηματοδοτικός φάκελος, όπου πρέπει να δούμε πραγματικά πόσους πόρους θα διαθέτουμε στην πράξη στα πλαίσια του φακέλου αυτού. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, άλλες παρατηρήσεις όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη. Έχουμε κερδίσει και χρόνο, θεωρώ. Ο κύριος Τρασκόφσκι είναι μαζί μας. Μάλιστα, εδώ είστε. Πολύ ωραία. Αν θέλετε να έρθετε λίγο πιο κοντά εδώ πέρα, μπορείτε να φέρετε και την κάρτα σας μαζί σας. Προτιμάτε να μείνετε πίσω, στα πίσω έδρανα μάλιστα. sorry. would just, uh, I just welcome uh, Mrs. our first Vice President. Κύριε Πετικάινεν, η πρώτη μας αντιπρόεδρος είναι μαζί μας. Έχουμε και γνωμοδότηση από την ΙΤΡΕ. Ε, ο κύριος ε, Τσαρασκόφσκι λοιπόν είναι ο συντάκτης ε, γνωμοδότησης. Η κυρία Βάιλερ είναι σκιώδης, ο κύριος Χατζημαρκάκης δεν είναι εδώ μαζί μας. Ο κύριος Έγκστρομ, εγώ είμαι εδώ. Και η κυρία Ρούλε θα, θα μας καλύψει μάλιστα. Νομίζω ότι όλοι οι σκιώδεις ε, είναι εδώ. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο προφανώς μπορεί να το κάνει. Ο Ρίτσαρτ Σβέτον είναι εδώ. Ναι, είστε εδώ. Πολύ ωραία. Ο Ρίτσαρτ ε, Σουέταμ είναι εδώ από την DG Information Society. Κύριε Τρασκόφσκι, λοιπόν, ποια είναι η αποψή σα για την πρόταση αυτή. Παρουσιάστε μας την γνωμοδότησή σας, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά. Και εσείς γνωρίζετε αρκετά πράγματα όσον αφορά την περαιτέρω χρήση πληροφοριών, την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Θεωρώ ότι μπορούμε να δείξουμε θετική στάση, γιατί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλή. Ο συνήθω όμω, οι ευρωβουλευτέ καταφέρνουν να βρουν τρόπου βελτίωση του και αυτό ακριβώ πράξαμε κι εμεί. Αυτό έκανα μέσω τροπολογιών που πρότεινα. Το πιο σημαντικό είναι ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις, μάλλον προς τον τρόπο εργασίας, προς τον πρώτο λειτουργίας. Εμείς θέλουμε να έχουμε κάποιους καλύτερους ορισμούς, να είναι πιο ρητοί. Το πιο σημαντικό είναι το όλο εγχείρημα να μπορεί να λειτουργήσει υπέρ τη καινοτομία και τη οικονομική ανάπτυξη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όταν διανύουμε μια περίοδο κρίση. Πέντε σημεία θέλω να θίξω. Πρώτον, θα πρέπει κάποιοι ορισμοί να γίνουν λίγο πιο συγκεκριμένοι. Πρώτον, όσον αφορά τα μηχανοργανώσιμα μορφότυπα. Θέλουμε να είμαστε λίγο πιο σαφείς ως προς τον όρο αυτό. Θέλουμε από τεχνολογικής πλευράς να είναι ουδέτερο αυτό ο ορισμό και επιθυμούμε επίση να κρατήσουμε το μορφότυπο αυτό ώστε να τον πιο ανοιχτό και όσο πιο φιλικό προς το χρήστη. Γι' αυτό το λόγο προτιμούμε τους ανοιχτού μορφότυπους. Μπορούμε να αποδεχτούμε και άλλους μορφότυπους, αλλά μόνο κατ' εξαίρεση. Τασόμαστε σαφώς υπέρ των ανοιχτών μορφοτύπων, γιατί θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή για τον τελικό χρήστη. Δεύτερον, περιφθοριακό κόστος και εδώ πέρα θέλουμε να είναι πιο σαφής ορισμός. Θέλουμε εδώ πέρα να αναφερόμαστε μόνο στο κόστος το οποίο απαιτείται προκειμένου να υπάρχει επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Κατ' εξαίρεση πάλι μπορούμε να δεχθούμε άλλες διατάξεις, θα πρέπει όμως οι εξαιρέσεις αυτές να είναι ελάχιστες και περιορισμένες και να καθορίζονται εκ των προτέρων. Ανοιχτές άδειες τώρα, τρίτο ζήτημα. Αναφέρθηκα στο ζήτημα αυτό και στο παρελθόν. Αναφερόμαστε εδώ πέρα πάλι στο να είναι τα έγγραφα αυτά πιο διαθέσιμα. Θέλουμε ανοιχτέ άδειε προκειμένου τα έγγραφα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσο περι από τον περισσότερου χρήστε και θέλουμε να υπάρχει και μία τυποποίηση όσον αφορά των αδειών αυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αν θα ήταν καλύτερα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό σύστημα αδειών. Ένα ζήτημα το οποίο στο μέλλον πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέταρτον, ηλεκτρονικά μέσα. Θα θέλαμε η επαναχρησιμοποίηση και τα αιτήματα μεταχείρισης επεξεργασίας να γίνονται βάσει συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων. Γι' αυτό σβήσαμε και τον όρο «where appropriate» γιατί τα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να αποτελούν το εφαλτήριο, το σημείο κίνησης. Αν πραγματικά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό προς το συμφέρον της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιείται, ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιείται όσο το περισσότερο. Πέμπτο, εποπτεία, παρακολούθηση. Το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε η συζήτηση που κάναμε για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο το ζήτημα αυτό. πολλοί, ακόμα και στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, θέλουν να δημιουργήσουν νέε αρχέ, νέε οργανώσει. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα αυτό. Α μην δημιουργήσουμε νέε οντότητε, νέε αρχέ, α χρησιμοποιήσουμε τι υφιστάμενε εποπτικέ αρχέ, οι οποίε θα κληθούν να παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία. Όσον αφορά επίση τι απαιτήσει υποβολή αναφορών, θα θέλαμε να γίνουν λίγο πιο ρεαλιστικέ. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι οι απαιτήσει υποβολή αναφορών θα πρέπει να αφορούν τριετή περίοδο και όχι ετήσια περίοδο και αλλάξουμε επίση και την γλώσσα, τη διατύπωση, όπου λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν αναφορές όσον αφορά την ε, διαθεσιμότητα των ε, δεδομένων, των πληροφοριών και όχι το επίπεδο χρησιμοποίησής τους ή επαναχρησιμοποίησής τους. Θέλουμε να είμαστε όσο τον πιο ρεαλιστικοί. Θέλουμε υποβολή αναφορών, θέλουμε να γίνεται μια εποπτεία. Α γίνει από τι εφιστάμενε αρχέ όμω και α γίνει η εποπτεία αυτή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην λειτουργεί εναντίον των κρατών μελών, να μην δημιουργεί ουσιαστικά περαιτέρω γραφειοκρατικό άκθο για τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης ηγητές για την εξαιρετική συνεργασία, να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Κόμη, η οποία δέχτηκε να αλλάξει η σειρά στη μερίσια διάταξη, προκειμένου να σας μιλήσω εγώ σήμερα, γιατί δεν θα είμαι παρόν αύριο. Ευχαριστώ. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Κυρία Κοράτσα μου. Ευχαριστώ πολύ. Uh, right. Um... Thank you very much indeed for uh, picking up a number of points which also came up. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ και τον εισηγητή που ήρθε νωρίτερα. Ε, να ακούσουμε τους και εισηγητές και όποιον άλλον θέλει να μιλήσει. Η κυρία Βάιλερ πρώτη και μετά ο κύριος Χατζημαρκάκης, ο κύριος Έγκστρομ που κατέφθασε και εγώ και η κυρία Ρούλε. Πάμε. Mr. Engstrom is, is the shadow for this. But if uh, Mrs. also wants to contribute, you can. No, no, no, no, no. Are oh, you the shadow for it? All right, sorry. Are uh, you, I'm uh, Mr. Engstrom Λοιπόν, ποιο θα μιλήσει από εσά, ο κύριο Engstrom, η κυρία Ρούλε, αποφασίστε. Λοιπόν, αλλά πρώτα η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσασκόφσκι. Χαίρομαι πολύ που αλλάξαμε τη σειρά και το συζητούμε σήμερα το θέμα σας. Την έκθεσή σας αυτή την έχουμε ξανασυζητήσει ε, και την ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πιστεύω ότι με τις τροπολογίες τώρα βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε επιφυλάξει σχεδόν καθόλου την εξισμία, μία, να σας την αναφέρω. Στην εισαγωγή σας, κυρίως αναφέρεστε στη σημασία ε, όλων αυτών για την οικονομία και για τις επιχειρήσεις. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, ένας άλλος κύκλος χρηστών που είναι οι πολίτες βεβαίως αλλά και οι δημοσιογράφοι όσο και οι επιστήμονες που μας ενδιαφέρει και εμάς αυτό είναι ένα βρύφασμα ενδιαφερομένων και καλά κάνει και σωστό είναι αυτό και κατά την άποψή μας ε, ορθότατο ένα δεύτερο για το περιθωριακό κόστος και γι' αυτό συμφωνούμε είπατε ότι θα πρέπει να είναι ε, καλά τεκμηριωμένο και συμφωνώ και ε, ελέγξιμο. Δηλαδή, ε, δεν είναι μια τυχαία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα κράτη-μέλη πολύ διαφορετικά κινούμαστε. Στη Σκανδιναβία και σε κάποιες άλλες βόρειες χώρες υπάρχει άλλη φιλοσοφία, όπου αυτό είναι αυτονόητο. Και σε κάποιες χώρες μεταξύ αυτών και δική μου, είναι τεράστιες οι δυσκολίες να το παραδεχθούν. Εξού και η πρωτοβουλία αυτή με τη φιλοσοφία ότι η πληροφορία θα πρέπει να είναι για τους πολίτες. Είπα και την περασμένη φορά στη συζήτηση ότι λυπάμαι που ο επόπτης προσωπικών δεδομένων δεν συμπεριλήφθη στην προσπάθεια αυτή, εκ των προτέρων μάλιστα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κύριε Σίγητα ε, πώς θα γίνει αυτό στην τελική φάση ε, και ε, διατύπωση πρέπει να συμμετέχει από τις προστασίες δεδομένων. Να το γράψουμε δηλαδή ότι θα συμμετέχει εκ των προτέρων στις διαβουλεύσεις. Επίσης θεωρώ σημαντικό και σωστό το γεγονός ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε νέα υπηρεσία, αλλά να παραμείνει στη διοίκηση αλλά θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό γιατί μέχρι σήμερα εκεί που δεν υπήρχε καλή πρόσβαση στην πληροφορία αυτοί που μπλόκαραν ήταν πολύ συχνά οι κρατικές αρχές. Εάν τώρα τους αναθέσουμε να ε, διευθετήσουν και αυτό το θέμα, δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να τον μπλοκάρουν, αλλά να καταλάβουν την ίδια τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας και να την εφαρμόσουν. Και κάτι άλλο, δεν ξέρω πού πρέπει να το γράψουμε αυτό, ε, σε περίπτωση που δεν λειτουργούν αυτά καλά υπάρχει και ο διαμεσολαβητής και ο εθνικός και ο ευρωπαίος διαμεσολαβητής που φροντίζει να μην ε, αποσιωπώνται οι πληροφορίες αυτές και να φτάνουν στον τελικό τους ε, αποδέκτη που μπορεί να είναι πολίτες, ή δημοσιογράφοι κτλ. Και χαίρομαι που μιλάτε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ε, προσωπικής ζωής. Το υποστηρίζω πάρα πολύ γιατί σήμερα ούτε αυτό είναι πλέον αυτονόητο και καλό να το γράφουμε. Γενικότερα λοιπόν είναι μια προσέγγιση καλή, ρεαλιστική και ας ελπίσουμε να αξιοποιηθεί και με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν εντάξει. Ήδη από γεννησιμιού της. Το είπε και η κυρία Βάιλερ. Ο εισηγητής θα βελτίωσε με τους ορισμούς και συγχαρητήρια. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την κυρία Βάιλε. Ωστόσο, στα κράτη-μέλη παραμένουν πολύ μεγάλες διαφορές. Το διαπιστώνει και ο ίδιος ο εισηγητής. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν την οδηγία πλήρως και σωστά. Γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλοί αποκλειστικές ε, ερμηνείες και ρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ακριβώς το δημόσιο, για την επαναχρησιμοποίηση των ίδιων τους ε, των εγγράφων ή ε, εγγράφων άλλων χρηστών ε, που προχωρούν σε επαναχρησιμοποίηση, reusers όπως λέγονται. Επίσης, οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι και πιο φθηνές ε, διαδικασίες για τη διευθέτηση ε, και επίλυση διαφορών και διενέξεων. Και αυτό το έχει υπόψη του εισηγητής και το λέει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, Mrs. Η κυρία Ρούλε, συμφωνώ και με τις ευχαριστήσεις και με τους επένους. Είχαμε ήδη μια προηγούμενη καλή συζήτηση και ο εισηγητής μας παρουσίασε τις βασικές του ιδέες. Ήδη από τότε θεώρησα ότι είχε τη σωστή προσέγγιση. Τώρα το έχει μεταφέρει αυτό το πνεύμα και στις ε, τροπολογίες του. Συμφωνώ απολύτως ότι η προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων είναι ικανοποιητική, ας πούμε στην τροπολογία 13 τα λέει θαυμάσια ή και σε μια άλλη τροπολογία η 6 νομίζω είναι, τα ξεκαθαρίζει αυτά. Και μένα ε, με απασχολεί πολύ και το θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμο ότι αλλάξατε και ορίσατε σαφώς το θέμα των τελών που καταβάλει κανείς στην τροπολογία υπαριθμών 10. Οπότε εγώ δεν χρειάζεται να κάνω καθόλου τροπολογίες ούτε η ομάδα μου πιστεύω. Ε, μπράβο, καλή δουλειά και καλή επιτυχία. Uh, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις ως σκιώδης εισηγητής για την πρόταση αυτή και είχα εργαστεί και στην αρχική πρόταση όταν πήγε στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Ξεχνάμε ορισμένες φορές το ότι ήταν πραγματικά καινοτόμη πρόταση αυτή όταν πρώτο προτάθηκε και ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα μία εξελιγμένη της εκδοχή. Δεν ξέρω πόσες πληροφορίες καταφέραμε να συλλέξουμε, πάντως είμαι σίγουρος ότι η πρόταση αυτή πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική πρόοδο να αφορά την επανεχρησιμοποίηση των πληροφοριών, ένα σύστημα το οποίο μπορεί να, οδηγεί, να λειτουργήσει προς το συμφέρον της κοινωνίας και της ψηφιακής οικονομίας. Έθεσα το ρώτημα την προηγούμενη φορά, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να εμπλέξουμε περισσότερο και κάποιους δημόσιους οργανισμούς που κάνουν ένα πολιτιστικό έργο, πολιτιστικούς οργανισμούς ουσιαστικά. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια ευελιξία όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Θα πρέπει βέβαια να καταφέρουμε να δούμε και ποια θα είναι τα λειτουργικά έξοδα των οργανισμών αυτών. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί και ας μην επιβάλλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σύστημα το οποίο θα είναι πάρα πολύ αυστηρό προς την τιμολόγηση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε τέλος θα θεσπίζεται δεν θα είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε τελικά να εμποδίζει τη διάχυση αυτών των δεδομένων. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός ε, εποπτείας και είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιβάλλει κάποιο άκαμπτο σύστημα, αλλά δίνει κάποιες καθοδηγήσεις, κάποιες ενδείξεις. Εδώ πέρα μάλιστα ερχόμαστε σε αντίθεση με άλλες προτάσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τις δημόσιες συμβάσεις, όπου το σύστημα το οποίο προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ πιο άκαμπτο. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Γενική Διεύθυνση Information Society που έχει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο φάκελο αυτό. Οι ε, τροπολογίες του συντάκτη γνωμοδότησης αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα. Θα εξετάσουμε πάντως εκ νέου το κείμενο για να δούμε αν θα πρέπει να έχουμε βελτιώσεις μέσω επιπλέον τροπολογιών. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ουδής. Να δώσω το λόγο στον Ρίτσα Σουέτεναμ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τον ακούσουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί έχει μεγάλη εμπειρία στο τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω είναι μια στιγμή ιδιαίτερη ε, ικανοποίηση για τον Επίτροπο το να βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια ομοφωνία ως προς την πρόταση της Επιτροπής. Βεβαίως έχετε δίκιο αρχικά δεν ήταν κάτι που θεωρήθηκε από την Επιτροπή ιδιαίτερη προτεραιότητα. Βεβαίως έγινε το πρώτο βήμα από το Κοινοβούλιο, τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ένα δεύτερο περαιτέρω βήμα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα Παραμένει η αρχική ιδέα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και από άλλους. Άκουσα ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να υποβληθεί για νομοδότηση στον φορέα προστασία των δεδομένων. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει δυναμικό στον τομέα αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν προσωπικά δεδομένα. Και για το λόγο αυτό ακριβώς η, συγκεκριμένη οδηγία το αποκλεί αυτό από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Και βεβαίως η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα για το πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είμαστε υπέρ των προτάσεων διατύπωσης που στόχο έχουν να υπογραμμίσουν το συγκεκριμένο σημείο. Το Κοινοβούλιο έχει, ασχολείται με την πρόταση που έχει υποβληθεί από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει την ενιαία εφαρμογή των κανόνων αυτών που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Νομίζω ότι είναι η πιο κατ κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν κανόνες. Και είναι καλό όλα αυτά τα δεδομένα, που, ε, τα στοιχεία που αφορούν την προστασία των δεδομένων να συγκεντρωθούν σε ένα και μοναδικό σημείο. Διαφορετικά δημιουργείται πολύ μεγάλη σύγχυση. Ας επικαιροποιήσουμε τους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες αυτές. Δεν θα πρέπει αυτή η νομοθεσία να επηρεάσει τους ε, τα προβλεπόμενα για την προστασία των δεδομένων και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα όπου εφαρμόζονται. Ωραία, σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω τα όσα είπατε σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να ενδιαφέρει εδώ. Νομίζω ότι είναι καλό το ότι κινούνται αυτά τα δύο σημεία παράλληλα. Ορισμένα δεδομένα θεωρούνται προσωπικά, ενώ σε άλλες χώρες όχι, δεδομένα που αφορούν τον ε, δημόσιο τομέα. Ας πούμε, οι αριθμοί κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ενδεχομένως, κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο θέλει να ελέγξει την ε, προέλευσή του και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για το πληροφορηθεί. Σε ορισμένες ε, χώρες αυτά τα ε, στοιχεία θεωρούνται δεδομένο ο αριθμός κυκλοφορίας. Βεβαίως γίνονται προσωπικά όταν συνδέονται με το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλα θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των χωρών. Και θα πρέπει να δούμε εάν είναι πληροφορίες ε, ε, που ε, είναι γενικού ειδικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να δούμε για τι στοιχεία μιλάμε. Μιλάμε για φωτογραφίες των σπιτιών, των κατόχων. Ίσως αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Κύριε Στασκόφσκι, τι θέλετε, ε, να κάνετε μία ανακεφαλαίωση. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, όπως το θέμα της ιδιωτικότητας ή της ε, φύσης των πληροφοριών. Γι' αυτό το λόγο υποβάλαμε τροπολογίες. Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει γνωμοδότηση των ε, φιλελεύθερων ε, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα, μια ιδέα για το πόσο θα μπορούσαμε να επιληφθούμε αυτών των θεμάτων. Κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Κοίταξτε, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που είναι ένα θέμα που αναφέραμε σε, όλα, σε όλες ε, τις τροπολογίες, σε γενικές γραμμές, όλα αυτά είναι υπέρ των πολιτών. Σε ό,τι, Ω προς το θέμα της εποπτείας, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε φορείς ενδεχομένως, όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποια ε, τροπολογία σε ό,τι αφορά το ρόλο του ομπούτσμανα. Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί. Σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά, τους πολιτιστικούς φορείς ή το ε, οριακό κόστος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς εννοούμε εδώ. Σε τι κίνδυνο αναφερόμαστε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας, περιμένω τις ε, τροπολογίες σας και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε σύντομα με τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού. Για μία ακόμα φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, 29 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι είναι η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες αυτές στην συνεδρίαση μας στις 10 Ιουλίου. Θα εξετάσουμε συμβαστικές τροπολογίες στις 17 Σεπτεμβρίου, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 18 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία στην Ήτρα θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν κάποιο χρόνο, θα έχουμε και χρόνο λίγο αργότερα να ενσωματώσουμε στι βασικέ τροπολογίε και τροπολογίε που ενδεχομένω να υποβληθούν κάποια στιγμή αργότερα. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κερδίσει πέντε λεπτά μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω αν είμαστε όλοι στην αίθουσα, γιατί ορισμένε φορέ οι σκιώδει ηγητέ φτάνουν τελευταία στιγμή. Ο κύριο Φάμπε μου είπε ότι θα αντικαταστήσει κάποιον σκιώδη ηγητή. Ο κύριος Σμίτ είναι εδώ, ο κύριος Έγκστρομ επίσης, ο κύριος Μπίλανο απουσιάζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται, ο κύριος Χάινεν είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχεδόν απαρτία λοιπόν έχουμε κύριε Κοφεράτη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Μάλιστα θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότης του κυρίου Κοφεράτη για την πράσινη βίβλο προς μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων πριν από μερικές εβδομάδες. Ακούσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Κοφεράτη για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησή του και θα ακούσουμε έπειτα και τους πιο ηγητές και οποιονδήποτε άλλο θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, όπως είπα και προηγουμένως, όταν είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας, αυτό που υπογράμισε υπογραμμίστηκε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του, αλλά και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ορισμένων ανετικών φαινομένων που αφορούν όλες τις χώρες της, Ευρωπα... της Ένωσης. Για παράδειγμα, σκέφτομαι πως η πληρωμή, η ηλεκτρονική πληρωμή θα μπορούσε να βοηθήσει την καταπολέμηση της γκρίζας ε, της παραοικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των φορολογικών απατών. Συνεπώς η ανάγκη να, να γίνουν ενιαίοι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντική. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και για το λόγο αυτό μετά από διαβουλεύσεις προσπάθησα να συμπεριλάβω στο κείμενο ορισμένα σημεία που αντικειμενικά μου φαίνονται πιο σημαντικά και ενδεχομένως ε, δεν έχουν επιληθεί στο κείμενο της Επιτροπής. Απευθυνόμαστε στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής χρειάζεται ασφάλεια, χρειάζεται διαφάνεια και θα πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη μπροστά σε αυτά τα μέσα. Γιατί πρόκειται για μέσα τα οποία απαιτούν μία διαδικασία που δεν είναι πάντοτε μέρος της καθημερινής πρακτικής των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων πολιτών ή των πολιτών ε, που είναι ηλικιωμένοι ή που δεν είναι αρκετά μορφωμένοι. Για να κατακτήσουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη των πολιτών, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε σε όλους τους χρήστες σωστή πληροφόρηση. Πολύ συχνά οι χρήστες κατακλείζονται από ανώφελες πληροφορίες ή παραπλανητικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά την χρήση χρησιμότητα των ε, μέσων αυτών. Συνεπώς, σωστή πληροφόρηση και διαφάνεια. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε για να κατακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το δεύτερο βήμα αφορά την προάσπιση των συμφερόντων τους, των δικαιωμάτων τους. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δράσουμε με στόχο να ενισχύσουμε την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και σε επίπεδο τομικό και σε επίπεδο συλλογικό. Σε μία μετέπειτα φάση θα συζητήσουμε Ποιε θα μπορούσαν να είναι οι κατάλληλες μορφές για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει, θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι όταν χρησιμοποιούν αυτό το μέσο έχουν τη δυνατότητα να προφυλαχτούν από οποιαδήποτε αλλαγή είτε πρόκειται για πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών ε, που θα μπορούσε να προκύψει. Δηλαδή, ακόμα και η βεβαιότητα του νόμου, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είναι σημαντική για να μπορέσει κανείς να έχει την εξασφάλιση ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός χρηστών θα χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο πληρωμής και έτσι ώστε αυτός ο τρόπος πληρωμής να γίνει ένα αποτελεσματικό μέσο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ίδια τα μέσα, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια τυποποίηση. σε επίπεδο ευρωπαϊκό, που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια. Υπάρχουν συστήματα που παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Άλλα συστήματα που είναι λιγότερο ασφαλή. Υπάρχει διαφορά στη χρήση των διαφόρων ε, καρτών ε, υπάρχουν κάρτες που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς ένα δικό του κωδικό ή κάρτες που ενεργοποιούνται με μία ε, ε ένα μαγνητικό κωδικό. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους χρήστες, θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκά ε, πρότυπα και εδώ οι λύσεις θα μπορούσε να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Υπάρχουν συστήματα διπλής, διπλού ελέγχου που είναι ε, διπλής πιστοποίησης που είναι πιο αποτελεσματικά από τα άλλα. Το πρώτο σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι την τυποποίηση όλων των διαδικασιών σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Για να ευνοηθεί, για να προωθηθεί αυτή η τυποποίηση θα πρέπει να υπάρχει και μία διαφανής αγορά. Μία αγορά στην οποία δεν, δεν δημιουργούνται μονοπόλια. Γιατί ο κίνδυνος και εδώ, όπως και σε άλλες δραστηριότητες που είναι από την Επιτροπή, ε, υπάρχει ο καθοριστικός ρόλος των μονοπωλίων. Μερικές φορές ε, τα ε, μονοπόλια μπορούμε να τα καταλάβουμε με την πρώτη, άλλες φορές ε, είναι, βρίσκονται σε μια λανθάνουσα κατάσταση, αλλά επηρεάζουν τις ελεύθερες συναλλαγές και τελικά έχουν αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον τρόπο χρήσης αυτών των μέσων, αλλά και σε ό,τι αφορά το κόστος που έχουν. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δράσουμε και να έχουμε μία διάδοση των μέσων αυτών πληρωμής, αλλά παρέχοντας εγγυήσεις διαφάνειας και δυνατότητας ελέγχου από πλευράς όλων των χρηστών. Εκτός από αυτό, οι υπηρεσίες πληρωμών θα, θα πρέπει να γνωρίζουν εάν αυτός που κάνει την πληρωμή είναι σε θέση να καταβάλει τα χρήματα. Δεν είναι θέμα παραβίασης της ιδιωτικότητας, δεν είναι θέμα πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα. Απλά και μόνο θα πρέπει να υπάρχει μία επιβεβαίωση που αφορά το αξιόχρεο, τη φερεγγιότητα του ατόμου που χρησιμοποιεί αυτό το μέσο για να αποφευθούν διαφορές και για να, αποφευθεί, ε, να αποφευθούν και οι απάτες. Τέλος, υπάρχει το πρόβλημα του κόστους αυτής της ε, δραστηριότητας. Πιστεύω ότι το πρώτο βήμα αφορά την εναρμόνιση των προμηθειών που διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη και σε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε μία κατάργηση του κόστους, του υπάρχοντος κόστους σήμερα η άμεση εξάλληψη, η άμεση κατάργηση ενδεχομένως είναι αδύνατη. Και κατά κάποιο τρόπο είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε σε δύο φάσεις. Ε, η πρώτη αφορά την εναρμόνιση, η οποία ευθύ εξ αρχής είχε στόχο την επίλυση του προβλήματος των προμηθειών, οι οποίες καταβάλλονται από το χρήστη. Δηλαδή προβλέπεται ένα τελικό σύστημα όπου το ποσό θα καταβάλλεται από τις ε, τράπεζες ή από τους χρηματοπιστωτικούς ε, οργανισμούς. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω αφορά την ανάγκη που υπάρχει να δοθεί, να διαδραματίσει κάποιο ρόλο η Επιτροπή και καθώς και η Κεντρική Τράπεζα για να ξεπεραστεί η ιδέα ότι η αυτορύθμιση είναι επαρκής. Χρειάζεται ένας τρόπος, ένα μέσο και χρειάζονται αυτοί που θα χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για να μπορούν να προβαίνουν σε έναν έλεγχο. Και είναι σημαντικό οι φορείς αυτοί να έχουν ένα σύστημα κοινοποίησης επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούν για να έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ποσοτικές αλλά και ποιοτικές αξιολογήσεις που αφορούν την όλη διαδικασία και τις ποσότητες που αφορά ως προς την χρήση των ε, ηλεκτρονικών πληρωμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Σέντο με τον οποίο είχα τη δυνατότητα Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνουν, θα μπορούσαν να καλυφθούν τα ορισμένα σημεία χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Είμαι στη διάθεσή σας στη διαθεσή σας για να εξετάσω τις ε, τροπολογίες που θα υποβληθούν. Μιλήσαμε ήδη για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω για τη συμβολή σας και μετά θα δούμε τι θα έπρεπε να κάνουμε τις τροπολογίες. Uh, uh, σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την ε, εργασία που κάνατε. Θεωρώ ότι ε, η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. 40 ερωτήσεις νομίζω ότι τίθενται. Κύριε Σβάμπ, μιλάτε εσείς ε, εξ ονόματος του κυρίου Αριάτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι με τον συνάδελφο Κοφεράτη, τον οποίο εκτιμώ εκπροσωπώ τον κύριο Παύλο Άριας που για οικογενειακούς λόγους χρειάστηκε να επιστρέψει ε, τελευταία στιγμή στην πατρίδα του. Πέρσι εγκρίθηκε η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε ε, αυτά τα θέματα για τις πληρωμές μέσω διαδικτύου για να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Και εκεί λέει ότι τα κράτη θα πρέπει να απαγορεύουν ε, στις ε, κάρτες και στις εταιρείες να χρεώνουν τους αγοραστές και τους καταναλωτές με επιπλέον κόστος, επιπλέον εκείνο που χρειάζεται πραγματικά. Ε, ας πούμε, όταν αγοράζει κανείς με πιστοτική κάρτα αεροπορικό εισιτήριο από το διαδίκτυο, πολλές φορές του ζητούν μία προμήθεια ή ένα καπέλο κοινός όταν πληρώνει με κάρτα. Δεν χρειάζεται όμως, πολλές φορές είναι άχρηστο αυτό το επιπλέον κόστο και χρειάζεται βελτίωση και χωράει και βελτίωση το ευρωπαϊκό σύστημα πλώμων. Γιατί αν συζητήσετε με εταιρείε που ε, δραστηριοποιούνται διασυνοριακά έχουν πολλά προβλήματα. όταν στέλνει κάτι με το ταχυδρομείο, είναι πολύ πιο ακριβώς στι διεθνεί μεταφορέ από τις εθνικέ, ακόμα και αν η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρότερη. Δεύτερο πρόβλημα η γλώσσα, τρίτον το νομικό πλαίσιο και τέταρτον ε, η πληρωμή και η διεκπαιρέωσή της. Ε, αυτά είναι τα τέσσερα λοιπόν προβλήματα που έχουν οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται ανά την Ευρώπη. Τα λέει και ο κύριος Κόφεράτη ε, και θα τα βάλει και στη γνωμοδότησή του. Ο συνάδελφος Άριας εργάζεται πάρα πολύ για την ψηφιακή εσωτερική αγορά και θα κάνει κάποιες τροπολογίες συμπληρωματικές ουσιαστικά που θα επικεντρώνονται στη σημασία και στις επιπτώσεις των επιγραμμικών πληρωμών ε, σε αυτή την ψηφιακή εσωτερική αγορά και στις εξελίξεις της. θα μιλήσει και για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών και ε, γιατί μπορεί να είναι θέματα αυτά συναφή. Και επίσης ε, ήθελα να πω ξανά, το είπα και την περασμένη φορά, ότι αυτό το σύστημα με τις πιστοτικές κάρτες, όλα τα συστήματα ε, βασίζονται στην εξή παραδοχή. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να έχουν πληροφορίες για ε, το, το, τη του ε, κατόχου της πιστοτικής κάρτας. Να ξέρουν αν μπορεί ο άνθρωπος να πληρώσει. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα διευρωπαϊκά ε, και διασυνοριακά. Χρειάζεται μια τυποποίηση, το είπε ο κύριος Κοφεράτη, αλλά ενδεχομένως και εκείνοι που χειρίζονται αυτά τα συστήματα θα πρέπει να επιληφθούν για να γίνει πιο απλή η διασυνοριακή συναλλαγή. Ε, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ε, που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Μια δυνατότητα είναι ε, τα πολύ τεχνικά ζητήματα αυτά, τα διαλειτουργικά, που είναι και πάρα πολύ ασφαλή. Και κοιτάω τον κύριο Άγκστρομ και εννοώ ασφαλή και ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τεχνικά μπορούν να μειωθούν οι νέες επενδύσεις εάν φροντίσουν οι εταιρείες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να λειτουργούν τα συστήματα τους. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για το ποιες ε, πληροφορίες διαβιβάζονται με ποιον τρόπο και πώς ε, όλο αυτό ε, προστατεύεται για να είναι δεδομένη η ασφάλεια στο διαδίκτυο και να έχουν όρεξη οι καταναλωτές γιατί θα είναι ασφαλείς οι αγορές τους να τις κάνουν και διαδικτυακά. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι εδώ τον κύριο Κοφεράτη. Uh, thank uh, Σας ευχαριστούμε, πολύ. Ο κύριος Σμίτ έχει το λόγο. Thank uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κοφεράτη. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα το οποίο συζητάμε και αυτό γιατί αφορά την ενιαία αγορά και το πώς θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τη σωστή της λειτουργία όπως είπατε και εσείς, έχει να κάνει με τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη το βασικό μας ζήτημα εδώ είναι ο καταναλωτής. Πρέπει να είναι φιλική η πρόταση προς τον καταναλωτή. Χρησιμοποιώ πολύ το διαδίκτυο, αγοράζω και πληρώνω στο διαδίκτυο και η εμπειρία μου είναι ότι γενικά λειτουργεί καλά αλλά παρόλα αυτά υφίστανται προβλήματα. Και νομίζω, κύριε Κοφεράτη, ότι έχετε καταφέρει να συμπεριλάβετε τα προβλήματα αυτά στην πρότασή σας. Επομένως, πολλές φορές βλέπουμε ότι όταν παραγγέλνει κανείς κάτι, αυτόματα και αμέσως, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, τα χρήματα φεύγουν από το λογαριασμό σας. Το προϊόν όμως, η υπηρεσία την οποία αγοράσετε, θα φτάσει μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα. Η λειτουργία πάντως αυτή, δηλαδή το ότι παίρνουν τα χρήματά σας αμέσως λειτουργεί πολύ καλά, αντίστοιχα θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε και ένα καλό επίπεδο ασφάλειας για τον καταναλωτή. Ο κύριος Έγκστρομ θα αναφερθεί φαντάζομαι σε κάποια ζητήματα ακεραιότητα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως να υπογραμμίσουμε τη διάσταση του καταναλωτή και ότι θα πρέπει πρώτα να είναι φιλική προς τον καταναλωτή και ότι θα πρέπει να μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τα οποία περιγράφονται εδώ. Και βέβαια ένα άλλο ζήτημα είναι η εμπιστοσύνη. Ορισμένες φορές θεωρώ ότι ο τρόπος που γίνονται αυτές οι πληρωμές αν λειτουργούν σφαιρικά σε παγκόσμιο επίπεδο, κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο επαφής... σε κάθε χώρα τουλάχιστον, έτσι ώστε αν εμφανιστούν προβλήματα, και εγώ ε, έχω συναντήσει πολλά προβλήματα, το όλο σύστημα είναι πολύ πολύπλοκο, είναι πολύ δύσκολο να έρθει στη συνέχεια κανείς σε επαφή με την επιχείρηση από την οποία αγοράζει κάτι. Θέλουν τα λεφτά μου, είναι έτοιμοι να τα πάρουν αμέσω, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσω στη συνέχεια με τι επιχείρησει αυτέ. Ορισμένε φορέ καλείται κανεί ακόμα και να τηλεφωνήσει στι Ηνωμένε Πολιτείε για να έρθει σε επαφή με την εν λόγω επιχείρηση και πολλέ φορέ δεν μπορώ να καταλάβω πώ λειτουργεί ακριβώ αυτό το σύστημα. Δεν είμαι πάντα υπέρ των εναρμονισμένων κανόνων και πάντα κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι το σχετικό. Κάτι που να προσεγγίζει την ευθυγράμμιση ακόμα και για τα τέλη, για το κόστος. Το είπατε κι εσείς αυτό. Έχω έρθει σε επαφή με ορισμένε επιχειρήσεις οι οποίες μου είπαν ότι σκοπεύουν να ακολουθήσουν κάποιους εναρμονισμένους κανόνες και μία διαφάνεια, ένα επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη και ενδεχομένως να απαγορεύσουν και κάποια τέλη. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει εδώ ένα περιθώριο ευελιξία το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να δράσουμε αναλογικά προφανώς και να πετύχουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Πολλές τροπολογίες επίσης θα ήθελα να υποβάλω και πιστεύω ότι ως συνήθως θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συνένεση, κύριε Κοφεράτη. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε αδιάλακτη στάση και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη διάσταση του καταναλωτή στην πρότασή σας. Και δεχομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο, λίγο παραπέρα όσον αφορά την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσβλέπω λοιπόν στις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Ξέρω ότι δεν πρέπει να κατανομάζουμε επιχειρήσεις, μόνο θα το θέλαμε πολλές φορές. Δεν πρόκειται πάντως να το πράξω. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έγκστρομ επόμενος. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και με τον προλαλήσαντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Όλο και περισσότερο ε, εξελισσόμαστε προς μια κοινωνία που θα χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές κάρτες και άλλες και πιστοτικές όλο και περισσότερο για τις πληρωμές και έτσι κι αλλιώς ε, συμβαίνει αυτό και θα πρέπει να ασχοληθούμε. Το πρώτο είναι αυτό που είπα και την περασμένη φορά που είχαμε ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίω και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ε, κανόνες αντικειμενικού και στεναρού που να λέγουν όταν ε, μια εταιρεία που εκδίδει πιστοτικές κάρτες αποκλείει μια εταιρεία, μια επιχείρηση από τη χρήση των καρτών της είναι πρόβλημα. Δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν τους κόψει την πιστοτική κάρτα και την πληρωμή από το διαδίκτυο, ε, αυτό σημαίνει το θάνατό τους για να κλείσουν το λουκέτο. Θα εξαφανιστεί η επιχείρηση αν δεν την αφήνει η εταιρεία που εκδίδει την πιστοτική κάρτα να πουλάει με πιστοτική κάρτα στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν παρευρίσκονται εδώ διάφοροι λόμπις από κάρτες και τέτοιους ε, παρόχους υπηρεσιών, αλλά είναι και προς το συμφέρον των ιδίων. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σκεφτεί κανείς μια κατάσταση όπου εκείνοι που εκδίδουν πιστοτικές κάρτες μπορεί να ε, πιεστούν πολιτικά ή διαφορετικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτρέψουν κάτι στην Ευρώπη και μια αντίστοιχη ή αντίθετη πίεση από το κοινό, την κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Δηλαδή πολύ γρήγορα μπορούν οι εταιρείε πιστοτικών καρτών να βρεθούν σε μία μέγενη. Αν όμως είναι οι κανόνες αντικειμενικοί, μπορούν να πούν και στους δύο ότι ναι, συμφωνώ μαζί σου, αλλά τι κρίμα, υπάρχει ο νόμος και με υποχρεώνει να τον ακολουθήσω και να συμμορφωθώ και ο κύριος Φαπ και ο κύριος Σμιτ ε, περιμένω από μένα να μιλήσω για την προστασία των δεδομένων. Θα το κάνω λοιπόν. Ε, στην ερώτηση 13 στην πράσινη βίβλο το έχασα ε, διαβάζοντας το θέμα. Ορίζεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς υπάρχουν διάφορες εταιρείες που δεν είναι τράπεζες και θέλουν πρόσβαση στα χρήματα που έχει κανείς στο λογαριασμό του όχι αν είναι φερέγγιος ναι ή όχι σε μία συναλλαγή, αλλά θέλουν το ακριβές ε, ποσόν να γνωρίζουν το καταθέσεων. Αυτό όμως είναι από τα πιο ευαίσθητα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Ίσως το πλέον ευαίσθητο, το τραπεζικό απόρριτο. Γιατί αν κάποια στιγμή αποδειχθεί ότι ο Α ή Β έχει πολλά λεφτά στην τράπεζα, πρώτον, θα κατακλειστεί από διαφημίσεις από την κάθε μεγάλη εταιρεία στον κόσμο, ε, θα είναι στόχος κάθε απατεώνα στον κόσμο ε, και όλοι θα απευθύνονται σε αυτούς για να τους αποσπάσουν χρήματα. Λοιπόν, ε, πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσουμε τους αυστηρούς κανόνες που έχουμε τώρα και να μην γίνει αυτό ένας φορέας διάδοσης της προφορίας για ε, το ύψος των καταθέσεων που έχει ο κόσμος γενικότερα. point on, on this. Ε, ε, άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω σχετικά. Α, για τα τέλη και τα λοιπά. Όταν ε, πρόκειται γενικά για τη ρύθμιση αυτού του συστήματος MIF, δεν ξέρω αν είναι ε, λογικό και σκόπιμο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Μπορεί να μην το κατάλαβα εγώ πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, επειδή δεν το έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τοποθετηθώ με σαφήνεια να σας πω αν είμαστε υπέρ ε, κατά ενός κανονισμού. Αυτά προς το παρόν σας ευχαριστώ. Α, ναι, και κάτι άλλο. Τροπολογίες θα κάνω φυσικά. Σε αυτές τις γραμμές που σας ανέφερα. Ο κύριος Μπιέλλαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα περισσότερα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε στην προηγούμενη μας συνεδρίαση όντως αντικατοπτρίζονται τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης οι πληρωμές στο διαδίκτυο και οι αγορές πληρωμών με κάρτα διαφέρουν πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Υπάρχει μια, ένα υπαρχει ενα διευκόλυνσης των πληρωμών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα όσον αφορά τα τέλη, θα πρέπει να είναι διαφανή και θα πρέπει επίσης και να μειωθούν και θα πρέπει να καταργηθούν εν τέλει. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό για μένα, γιατί στην Πολωνία δυστυχώς είναι αυθαίρετα τα τέλη αυτά και πολύ υψηλά και λειτουργούν εις βάρος των εμπόρων και των καταναλωτών. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που εντοπίζονται στην γνωμοδότηση, συμφωνώ με την κατεύθυνση γνωμοδότησης και θα την υποστηρίξω. Ήθελε και η κυρία Βάιλερ να μιλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους σκιώδης. Είναι σημαντικά αυτά που λέτε για τη διαφάνεια και οι προλαλήσαντες επίσης. Εγώ θέλω να πω ότι πολλοί καταναλωτές έχουν την εξής εμπειρία. Όταν θέλουν να εξοφλήσουν ένα λογαριασμό πιστοτικής κάρτας φεύγουν τα χρήματα από το λογαριασμό τους, αλλά περνάνε 5 και 7 ημέρες για να εξοφληθεί το ε, χρέος. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που πληρώνει ο καταναλωτής ε, αυτό δεν ε, αποδεικνύεται. Είναι σημαντικά αυτά για τους καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να μπορούν να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές πιστοτικές κάρτες. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και χρονική και σαφήνεια. Και εδώ μπαίνει το θέμα της διαφάνειας. Και η ασφάλεια είναι πάρα πολύ κρίσιμη και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ε, καθησυχαστούν ότι ε, γίνεται ασφαλής χρήση των δεδομένων τους. Πρόσφατα είδαμε πάρα πολύ ανησυχητικά φαινόμενα, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου και την ασφάλειά τους. Ευχαριστώ τον εισηγητή και προσβλέπω στην τελική μορφή της έκθεσης. Ευχαριστώ, κυρία Στάιλερ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Ασφα αναφέρθηκε σε το πολύ αυτό σημαντικό ζήτημα πώς διασυνδέεται η πρόταση αυτή με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στην οδηγία αυτή είχαμε αναφερθεί και στις ε, διασυνοριακές πληρωμές, καθώς επίσης και στα τέλη της προμήθειας που καλούνται να πληρώσουν πολλές φορές οι καταναλωτές που να αγοράζουν στο διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν στην πρόταση αυτή να ενσωματώσουμε κάποιες από τις παρατηρήσεις που είχαμε κάνει για την οδηγία και την προστασία των καταναλωτών. Θέλουμε σαφώς να δούμε πώς εξελίσσονται οι αγορές και στα πλαίσια της ψηφιακής αγοράς και να στείλουμε, αν θέλετε, όλες τις παρατηρήσεις αυτές στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων πρόκειται να ασχοληθεί με την πρόταση αυτή. Η έλλειψη διαφάνεια επίση είναι κάτι το οποίο μα απασχολεί καθώ επίση και το θέμα τη ανταγωνιστικότητα, το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ με την περιαγωγή, με τα τέλη περιαγωγή στην κινητή τηλεφωνία. Πολλέ φορέ εδώ πέρα τα πράγματα είναι χειρό, χειρότερα γιατί οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν καν ότι πληρώνουν κάποιε προμήθειε. Και κάτι ακόμα. Δεν χρησιμοποιούν όλε οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νόμισμα. Επομένω, οι διασυνοριακέ πληρωμέ πολλέ φορέ γίνονται με διαφορετικά νομίσματα. Και αυτό επηρεάζει βέβαια τα τέλη. Ο κύριος Κοφεράτη αναφέρθηκε στην βαθμία εξάλληψη όλων αυτών των τελών. Αν όμως προκύπτει κάποιο κόστος και αν πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις για να τονωθεί η αγορά αυτή, κάπου θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Επομένω, ακόμα και αν καταργηθούν τα τέλη αυτά, κάπου αλλού θα εμφανιστεί ένα άλλο κόστο. είτε στι ίδιε τι κάρτε, είτε ακόμα και στα τέλη των τραπεζικών λογαριασμών. Και όπω είπε και ο κύριο Σμιτ, δεν είμαστε εδώ πέρα για να επιβάλλουμε ένα επιχειρησιακό οικονομικό μοντέλο. Αυτό που θέλουμε είναι οι παράγοντε τη αγορά να μπορούν να λειτουργούν καλά. Αυτό ακριβώ είδαμε και στην περίπτωση του Ρόμινγκ, όπου οι παράγοντε τη αγορά δεν λειτουργούσαν προ το συμφέρον του καταναλωτή. Απαιτείται λοιπόν διαφάνεια για το τι ακριβώς πληρώνει ο καταναλωτής και για ποιο λόγο πρέπει να καταβάλουν τέλη, αν πρέπει να καταβάλουν τέλη. Και όταν απορροφούνται κάποια κόστη και κρηματοδοτούν κάποιες ενέργειες, πώς συμβάλλουν σε αυτά οι ε, καταναλωτές και τι ακριβώς γίνεται με διάφορες προσφορές, δίθεν προσφορές όπως τα δωρεάν κινητά τηλέφωνα, που στην πραγματικότητα δεν είναι κινητά και ουσιαστικά ο καταναλωτής τα έχει ήδη πληρώσει με έμεσους τρόπους. Νομίζω λοιπόν τα ζητήματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ιδιαίτερα ευαίσθητα και νομίζω ότι θα πρέπει να υποβληθούν με τον ένα τον άλλο τρόπο μέσω της γνωμοδότησής μας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε πολύ σωστά στα ερωτήματα αυτά τα οποία τίθενται. Έχουμε τον κύριο Χάινεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί μας. Ενδεχομένως ε, και αυτός θα ήθελε να μας διαφωτίσει για κάποια ζητήματα. Και ενδεχομένω θα καταφέρετε να ανταποκριθείτε και σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν θέσει οι συναδελφοί μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν γέννη θα έλεγα ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την γνωμοδότηση της Επιτροπής σας για την πράσινή μας βίβλο. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία με τους στόχους που έχουμε θέσει σε αυτή την πράσινη βίβλο. Το λαμβάνουμε λοιπόν αυτό υπόψη μας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μία συνένεση στο ότι ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε όλο και περισσότερο προς μια ψηφιακή αγορά ψηφιακών πληρωμών, ιδίω στα πλαίσια της ψηφιακής ενίας αγοράς. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο ανταγωνιστική αγορά πληρωμών στην Ευρώπη και γενικά μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο αποτελεσματικές οι αγορές αυτές από τις συμβατικές αγορές. Αυτό που ακούσαμε πολλές φορές είναι ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πρότασης αυτής. Αυτό ευθυγραμμίζεται και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις αρχές μα έγινε και μια δημόσια ακρόαση και αυτό ακριβώς είπαμε και εκεί. Αν δείτε τις μεθόδους πληρωμή που καλύπτονται από την πράσινη βίβλο, σε όλες τις περιπτώσεις ο τελικός χρήστη τελικά είναι ο καταναλωτή. επομένω αυτό διαφέρει με προηγούμενη νομοθεσία που είχαμε όσον αφορά διάφορα εμβάσματα, ή μεταφορές πληρωμών, όπου τότε αναφερόμασταν σε επιχειρήσεις. Αυτή τη φορά που μιλάμε για πληρωμές με κάρτα, μέσω διαδικτύου, μέσω κινητών τηλεφώνων, ουσιαστικά αναφερόμαστε στον καταναλωτή και από τη σκοπιά του τον καταναλωτή αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Αναφερθήκατε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας διαφάνειας, το ότι θα πρέπει να ενημερώνονται καταλήλως οι καταναλωτές, ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Πρέπει να σας πω ότι με την οδηγία των υπηρεσιών πληρωμής που εγκρίναμε πριν από μερικά χρόνια, έχουμε πλέον το απαραίτητο νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ασφάλεια των πληρωμών αυτών. Ουσιαστικά θα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομοθεσία αυτή στις νέες καινοτόμε πληρωμές που έχουν εμφανιστεί και την οποία αναφέρουμε στην Πράσινη Βίβλο. Επομένως αυτή η Πράσινη δίβλος και αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι δύο ζητήματα τα οποία συσχετίζονται άμεσα. Όσον αφορά τώρα την τυποποίηση, ιδίως σε σχέση με την ασφάλεια. Συμφωνούμε πλήρω με την παρατήρηση αυτή. όντω, ε, η ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ε, εκ των ουκ Θα πρέπει να διατηρήσουμε την προπόθεση αυτή σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία θα εγκρίνουμε για να δημιουργήσουμε μια πιο ανταγωνιστική αγορά. Η απέτηση, η προπόθεση τη ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική και να αναφερθώ και στο Secure Pay Forum, ένα σύστημα το οποίο έχει θεσπιστεί από τον ΟΣΑ και το οποίο δημιουργεί, θεσπίζει συγκεκριμένε προποθέσεις για ασφαλείς πληρωμές όσον αφορά τις πληρωμές που γίνονται στο διαδίκτυο, αλλά και άλλες μορφές πληρωμών αφορά το σύστημα αυτό. Και εμείς συμμετέχουμε στο φόρουμ αυτό, στις συζητήσεις που διοργανώνει αυτό το φόρουμ. Ο συντάκτης γνωμοδότησης αναφέρθηκε επίσης στα μονοπόλια. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο ότι θα πρέπει να αποφευχθούν τα μονοπόλια. Και αυτό αποτελεί βασικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τη πράσινη μας βίβλου. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ισότιμο επίπεδο δραστηριοποίηση διασυνοριακό για τις εφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και για τους νέους φορείς παροχής ηλεκτρονικών πληρωμών. Να μπορούν δηλαδή και αυτοί να μπουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αποτελεί ένα βασικό στόχο της πράσινης βίβλου. Να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο ανταγωνισμό, να δώσουμε περισσότερες επιλογές στον καταναλωτή και να έχουμε και πιο αποτελεσματικά, δηλαδή πιο οικονομικά μέσα πληρωμής για τους καταναλωτές. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των MIFs, των Interchange Fees, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ετέθη. Σαφώς χρειαζόμαστε και εδώ πέρα μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερη εναρμόνιση. Το εξετάζουμε αυτό με τους συναδέλφους μας από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο εκκρεμούν διάφορες υποθέσεις και προσφυγές όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε πρόσφατα στην υπόθεση της Mastercard για μια υπόθεση διαστοριακών πληρωμών και ήδη από το 2007 είχαμε πει ότι τα διασυνοριακά αυτά τέλη στις πληρωμές ήταν κατά τον ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις υποθέσεις αυτές που εκκρεμούν σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, όσον αφορά την διακυβέρνηση της ΕΠΑ των συστημάτων πληρωμών, συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε εκ των προτέρων δράση ιδίως όσον αφορά αυτούς που χαράσουν πολιτική. Έχουμε το Συμβούλιο ΣΕΠΑ και πέρυσι σε μία συνεδρίασή του προσπαθήσαμε να αναθεωρήσουμε το όλο σύστημα διακυβέρνησης ΣΕΠΑ και σύντομα θα υποβάλουμε, στο τέλος μάλιστα του έτους, μία πρόταση όσον αφορά τη διακυβέρνηση ΣΕΠΑ. Σε ένα εκτιμώντας μάλιστα του κανονισμού να φερόμαστε στο Συμβούλιο αυτό. Αυτό το οποίο θα εξετάσουμε είναι να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και πιο συγκεκριμένα πώς θα καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερο τους χρήστες στο σύστημα τυποποίηση το οποίο θα πρέπει να προκύψει. Υπάρχει λοιπόν ένας υψηλό βαθμός συνένεση για πάρα πολλά ζητήματα. Στα ζητήματα αυτά τα οποία έθιξε ο κύριος Κοφεράτη θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μα στην ανάλυση που κάνουμε. Έχει ε, ολοκληρωθεί και το σύστημα της δημόσιας διαβούλευσης. 300 περίπου απαντήσεις ε, λάβαμε, οι περισσότερες απαντήσεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν να λύσουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις και τις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλουμε ένα συνοπτικό έγγραφο στο οποίο θα συνοψίζουμε όλες αυτές τις απαντήσεις τις οποίες λάβαμε στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Και μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή δυνατόν θα προσπαθήσουμε να ανακοινώσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας αυτή. Κύριε Κοφεράτη, έχουμε περβεί το χρόνο που αναλογεί στην πρόταση αυτή, αλλά θα μπορούσατε ενδεχομένω να συνοψίσετε. Έχετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω. Ήθελα να σας πω ότι οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν θα ληφθούν σαφώς υπόψη. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω τους σιώδεις εισηγητές. Σε ό,τι αφορά θέματα ουσίας, θα ήθελα να πω τα εξής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη των τεχνολογιών. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο τροφοδοτείται από την τεχνολογία και που πάρα πολύ γρήγορα θεωρείται παροχημένο. Θα πρέπει να εστιαστούμε στην ανανέωση των τεχνολογιών. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τη χρήση των δεδομένων. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει να παρέχουμε εγγύσει για τα δικαιώματα των προσώπων, ξεκινάμε από το γεγονός ε, ξεκινάμε θεωρώντα δεδομένο ότι δεν πρέπει να ε, υπάρχει παραβίαση τη ιδιωτικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την ανταλλαγή, είναι μια σημαντική ανταλλαγή, αλλά πέρα από ένα συγκεκριμένο κατόφλι δεν θα πρέπει ποτέ να πάμε. Ενδεχομένω θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί στην εισαγωγή κάποιου καινοτόμου στοιχείου σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται εγγύσει για τον ανταγωνισμό. Αυτό το λέω ιδιαίτερα στον εκπρόσωπο τη επιτροπή που έκανε αυτή την παρατήρηση Υπάρχει ένα πρόβλημα σχέσεων με αυτό το χώρο των διάφορων φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα και των άλλων εμπλεκομένων. Θα πρέπει να μπουν σε ένα ίδιο επίπεδο έτσι ώστε η διαφάνεια να είναι το μέσο με το οποίο δημιουργούμε κίνητρα όχι μόνο για μια θετική προσέγγιση αλλά και για το σεβασμό των κανόνων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ευθύ εξ αρχή ότι τα άτομα που κινούνται σε αυτό τον ευρύτατο τομέα δυνητικής αγορά δεν έχουν την ίδια δύναμη. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών που είναι αδύναμοι. Ε, θα πρέπει λοιπόν στον τομέα αυτό να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να τους βοηθήσουμε. Good. thank you very much. It's been a useful debate. Ευχαριστώ πολύ χρήσιμη συζήτηση. Θα ήθελα μόνο να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει την Παρασκευή, την εξής πέμπτη διορθώνει ο Πρόεδρος, το μεσημέρι. Αλλά η Επιτροπή Οικονομικών θα ψηφίσει το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε τη σύνοψη των διαβουλεύσεων της Επιτροπής. Πάντως θα έχουμε πολλή δουλειά, μην ανησυχείτε. 10 Ιουλίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε εμείς 6 Σεπτεμβρίου. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε άλλη έκθεση του κύριου Κοφεράτη. Πολύ δουλειά έχει ο κύριος Κοφεράτη σήμερα το απόγευμα. Ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Είναι νομοδότηση για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και ο κύριος Φαπ πάλι είναι ε, υπηρεσιακός και οδησηγητής. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ε, είναι πάλι ο κύριος Σμιτ. Ποιος, κύριε Έγκστρομ, εσείς τι κάνετε εδώ. Πού είναι η κυρία Ρούιλε. Εδώ λέει η κυρία Ρούιλε ότι είναι σκιώδης γητρή. Είστε εσείς και ο κύριος Μπιέλαν. Ωραία. Παρακαλώ τον κύριο Κοφεράτη, αν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 5, θα σας είμαι ευγνώμων, αλλιώς θα φωνάζουν οι συντονιστές αλλά νομίζω έχουμε εδώ και τον κύριο Φίλιπ Σοντρέιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αρμόδια γενική Διεύρυνση. Δεν είμαι ε, σίγουρος ότι θα προλάβουμε να σας δώσουμε το λόγο, αλλά έχει το λόγο ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια γιατί είναι απαραίτητοι οι συντονιστές για την υγεία όλων μας. Ύστερα θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και αυτό βεβαίως κατά κάποιο τρόπο διευκολύνει το έργο μου. Σε ό,τι αφορά το θέμα και το κείμενο που υπευλήθη στην Επίτροπη, πιστεύω ότι λόγω των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθούμε στο θέμα των δικαιωμάτων των χρηστών. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε στις διάφορες αναφορές που κάνουμε και στους διάφορους ε, κανονισμούς που αφορούν το δίκτυο των υποδομών δεν θα πρέπει να συμπεριλάβονται, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι ε, υποδομές αλλά και οι άνθρωποι με σάρκα και οστά. Ε, πολλές φορές δεν γίνεται αυτή η διάκριση. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, να προσέξουμε τις πιο αδύναμες κατηγορίες. Άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ε, ε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, γιατί αυτό Τούτου του είδους ε, τα μέσα πάρα πολλές ε, φορές ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πάρα πολλούς ανθρώπους. Συνεπώς, ποιότητα στις παρεχόμενες επιχειρίες και υπηρεσίες και μέγιστη προσβασιμότητα στα πλέον αδύναμες κοινωνικές κατηγορίες. Θα πρέπει καταρχάς να γίνει μία εκ των προτέρων αξιολόγηση, δηλαδή στο σχεδιασμό των υποδομών ή στο σχεδιασμό των οχημάτων, είναι σημαντικό το θέμα της προσβασιμότητας να βρεθεί πριν από την κατασκευή της μεταφορικής υποδομής. Θα πρέπει να ε, απαιτήσουμε μέγιστη ασφάλεια και να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις έτσι ώστε η επίπτωση στο περιβάλλον να είναι πολύ περιορισμένη. Πάρα πολύ συχνά υπάρχουν αντιδράσεις, άλλες φορές χειραγωγούμενες, άλλες φορές αυθόρμητες ε, από πλευράς ε, μεγάλης μερίδας του πληθυσμού γιατί αμφισβητούνται ορισμένα ε, στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο έχουν ζήσει ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Από την αρχή λοιπόν θα πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός του περιβάλλοντος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε όλο αυτό το δίκτυο. Υπάρχουν ε, και ε, μερικές συγκεκριμένε πτυχές ε, που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Σκέφτομαι, ας πούμε, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σκέφτομαι και το θέμα των θαλάσσιων αυτοκινητόδρομων, ένα θέμα ιδιαίτερα καινοτόμο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το ε, λάβουμε υπόψη μας και να το... είναι ένα διατροπικό θέμα που ε, αφορά όλο το σύστημα των δικτύων. Υπάρχει ένα θέμα που δεν αφορά άμεσα εμάς. Δεν θα πρέπει όμως να αγνοούμε το θέμα των διαθέσιμων πόρων. Ήδη έχει γίνει ένα βήμα, αλλά πιστεύω ότι το δίκτυο έτσι όπως... Ε, διαμορφώνεται με τους υπάρχοντες πόρους δεν είναι εφικτό. Ενδεχομένως θα πρέπει να, να αναφερθούμε στο τι θα μπορούσε να γίνει. Σκέφτομαι τους ιδίους ε, πόρους που, που θα απασχολήσει το Κοινοβούλιο. Οι συντονιστές κατά την άποψή μου δεν μπορούν να παίξουν απλό διαχειριστικό ρόλο και να αφορούν τη διασύνδεση των διαφόρων τμήματων του δικτύου. Οι συντονιστές θα πρέπει να αποκτήσουν μια πολιτική σε εισαγωγικά εξουσία συνομιλίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τον προγραμματισμό και για την ε, κατασκευή των τμήματων αυτών του δικτύου. Ε, γιατί εάν ε, θα μπορούσαν να παρέμβουν εκ των προτέρων, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην εφαρμογή του συστήματος των μεταφορών ε, και γενικά και ειδικά θα μπορούσε να έχει επιληθεί. Είπα βεβαίως ότι πολλά από αυτά τα θέματα θα μπορούσαμε να τα επενεξετάσουμε και λέγοντας αυτό να σταματήσω σε αυτό το σημείο. Uh, Mr. Κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη πάλι για τα λεγόμενά του και να το συγχαρώ και εξ ονόματος και κατ' εντολήν της συναδέλφου Ιβάνοβα αυτή τη φορά ε, που δυστυχώς κολλείεται για αυτή σήμερα. Θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Κοφεράτη είναι προσανατολισμένος προς το χρήστη και για να το πω για την Επιτροπή μας προσανατολισμένος στον καταναλωτή στη γνωμοδότησή του. Για τη συνάδελφο Ιβάνοβα είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την πρόσβαση του πληθυσμού ολόκληρου σε τέτοια μέσα μεταφοράς που κυκλοφορούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δηλαδή και ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες αλλά και με περιορισμένη κινητικότητα να μπορούν να κυκλοφορούν. Αυτοί οι μεγάλοι άξονες ε, μεταφορών θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από όλους τους πολίτες της Ένωσης. Ε, επιπλέον, θα πρέπει η υποδομή να διευρυνθεί σε σημεία που θεωρούνται κόμβοι και αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο το δίκτυο και οι υποδομές και οι δυνατότητες συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα κυρία Ιβάνοβα τονίζει την οδική ασφάλεια που τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική αλλά και αυτό το λέει ο κύριος Σκοφεράτη ρητά. Τρίτον, αυτό που έχει σημασία είναι οι κυκλοφοριακοί αυτοί άξονες να αποφασιστούν ε, σε επικοδημητικό διάλογο. Και το λέω ε, ε, γιατί προέρχομαι από μια περιφέρεια που φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό μετά από μεγάλη δημόσια συζήτηση, μετά από τοπικό δημοψήφισμα ε, και πραγματικά τελικά ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από ό,τι αναφέρει ο τύπος για το σταθμό αυτό. Λοιπόν, ε, θα είναι σημαντική η συμμετοχή των πολιτών σε τέτοια έργα κατά την εκπόνησή τους και ευχαριστούμε και τον κύριο Κοφεράτη που τα λέει αυτά στην γνωμοδότηση. Πολύ λίγα σημεία μόνο που θέλουμε να τονιστούν περισσότερο, ε, οι άξονε των διευρωπαϊκών δικτύων σε διάφορους τομείς μεταφορών θα πρέπει να είναι ποιοτική εμπειρία για τους πολίτες ε, και όχι υπερβολικά δαπανηρή ταυτόχρονα. Άρα οι διοικητικέ απαιτήσει δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά ε, υψηλές να μπορούν, επαναλαμβάνω, όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση παντού στην Ευρώπη και όταν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε διάφορα κράτη-μέλη συγκεκριμένα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Παράδειγμα, αραιοκατοικημένες περιοχές που δεν υπάρχουν εναλλακτικές μορφές και εναλλακτικά δίκτυα οδικά ή άλλα. Οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτομίε θα πρέπει να αξιοποιούνται, λέει η κυρία Ιβάνοβα, έτσι ώστε να έχουμε τις πιο αποτελεσματικές και τις πιο φτηνές λύσεις για όλους τους πολίτες. Με καλή ενημέρωση για τις διασυνδέσεις, για τις ανταποκρίσεις και για τη μετάβαση από το ένα μέσο συγκοινωνιών μεταφορών στο άλλο στις συνδυασμένες μεταφορές. Και ένα πολύ πρακτικό ε, για να χρησιμοποιεί κανείς αυτούς τους άξονες θα πρέπει ο σημερινός κανονισμός να περιλαμβάνει και άλλες προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, σε μια πλατφόρμα ε, Ευρωπαίων χρηστών αυτών το μέσο μεταφοράς κοινώς επιβατών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Κοφεράτη και πιστεύω και εδώ ότι θα καταλήξουμε σε καλές λύσεις από κοινού πάντα. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σμιτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Γιατί άλλωστε κάναμε τη συζήτηση αυτή πριν από μερικές εβδομάδες και νομίζω, κύριε Κοφεράτη, ότι έχετε όντως ενσωματώσει κάποιες από τις παρατηρήσεις μας στην πρότασή σας. Και θα ήθελα να αφαιρθώ ιδιαίτερα στις τροπολογίες 2 και 30, που έχουν να κάνουν με το ρόλο των συντονιστών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός. Νομίζω ότι ε, αναφέρθηκα στο ότι ασχολούμαι με το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο αυτό στην πατρίδα μου και οποιοδήποτε το έχει πράξει αυτό ουσιαστικά γνωρίζει πόσο πολύπλοκα είναι τα πράγματα όταν πρέπει κανεί να δημιουργήσει ένα λιμένα, ένα δρόμο, ένα σιδηρόδρομο. Γιατί τελικά βρίσκεται αντιμέτωπο κανεί με όλου αυτού οι οποίοι παραπονιούνται. Όλοι θέλουν ένα σιδηρόδρομο, όλοι θέλουν στερεοδρομικέ γραμμέ, αλλά όχι δίπλα στο σπίτι του. Κάπου αλλού, κάπου μακριά. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ο συντονισμός ανάμεσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Προερχόμενος από μια αεροκατοικημένη χώρα σαν τη δική μου, θα έλεγα ότι το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στα διασυνοριακά ζητήματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, τα διάφορα κενά που υπάρχουν στι διαφορέ χώρε, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα κυκλοφοριακή συμφόρηση. Διαφορετικά θα καταλήξουμε με πάρα πολύ καλά διασυνοριακά συστήματα, αλλά το σύστημα θα χωλαίνει πάρα πολύ σε εθνικό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κάποια συνέπεια στο σύστημα το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας και νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα είναι όντως πολύ σημαντική και αν δεν καταφέρουμε να έχουμε τα νομικά μέσα, τότε θα πρέπει να δώσουμε στους συντονιστές μας όλο το απαραίτητο αυτό υποστηρικτικό προσωπικό, που θα τους επιτρέψει να επιτελέσουν αποτελεσματικά την εργασία τους και τελικά που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν μια πιο συντονισμένη αντιμετώπιση του ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει και από τους πολιτικούς μας σε εθνικό επίπεδο να τους ζητήσουμε να επηρεάσουν τους εθνικούς βουλευτές ή τους βουλευτές στα περιφερειακά κοινοβούλια. Διαφορετικά το όλο σύστημα το οποίο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να ολοποιηθεί στην πράξη. Αυτά έχω να σας πω κύριε Κοφεράτη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σμίτ. Ο κύριος Μπίελαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τις μεταφορές θα βοηθήσουν όχι μόνο τις ε, περιφέρειες στις οποίες ε, δημιουργούνται τα έργα αυτά, αλλά θα συμβάλλουν γενικότερα στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα νέα έργα με θα πρέπει πραγματικά να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι επιβάτες, οι χρήστες και θα πρέπει βέβαια να γίνουν και διαφανείς κοινωνικές διαβουλεύσεις. Θα ήθελα, έχοντας διαβάσει τις τροπολογίες, να τις σχολιάσω, αν γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα όσα λέγονται για τις διαβουλεύσεις με τον τοπικό πληθυσμό. Υποστηρίζω τις τροπολογίες 2 και 28. Πρέπει να σας πω επίσης ότι οι διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και πάντα να έχουν ως στόχο να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Θα πρέπει να αποφύγουμε καταστάσεις όπου έχουμε κάποιες τοπικές κοινότητες οι οποίες διαφωνούν παντελώς με κάποιο προβλεπόμενο έργο θα πρέπει ένα εγκεκριμένο έργο να έχει την ε, πρώτερη έγκριση της, ε, του τοπικού πληθυσμού. Θα προτιμούσα όσον αφορά την ανάλυση την οποία γίνεται, την γνωμοδότηση η οποία απαιτείται, να χρησιμοποιήσουμε την αρχική διατύπωση που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα και ότι θα πρέπει, όχι θα πρέπει να επιβάλλεται. Όσον αφορά την τροπολογία 8, ότι θα πρέπει να περιορίσετε στο ελάχιστο περιβαλλοντική επίπτωση, δεν είμαι πεπισμένο για την διατύπωση που χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μειώνουμε την αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον. Πέρα από αυτά δεν έχω να κάνω άλλες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Ενδεχομένως να μπορούσαμε να δώσουμε και δύο-τρία λεπτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος ε, Σαντχέν θα ήθελε να πάρει το λόγο και μετά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοφεράτη. Ευχαριστώ, μπορεί να, μπορεί να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Νομίζω ότι μπορούσαμε να, να καλωσορίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Κοφεράτη. Τονίζει μερικά σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μας, το θέμα της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, προσβασιμότητας. Επίσης, τονίζει το θέμα των συντονιστών και αυτό είναι ένα θέμα που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Σήμερα γίνεται μία συνάντηση των συντονιστών που θα συζητήσουν το θέμα της καλύτερης διάρθρωσης του διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες για να μπορέσουν να αποφευκθούν προβλήματα όταν τεθεί το θέμα της εφαρμογής του δικτύου ή της ανάπτυξης του δικτύου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τα άρθρα για την προστασία των περιβάλλοντος και την προβασιμότητα τα 42 και 43 έχουν ενισχυθεί όπως θα γνωρίζετε στην, στο Συμβούλιο το Μάρτιο διέγραψε αυτά τα άρθρα και έκανε μια απλή αναφορά σε αυτά τα θέματα στο εκτιμώντας προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Επιτροπής. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο μας υποστηρίζει και ελπίζουμε ότι πάνω σε αυτή τη βάση θα μπορέσουν τα άρθρα αυτά να ενσωματωθούν στον τελικό κανονισμό. Τελευταίο σημείο. Όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Σουάπ, θα πρέπει να αποφύγουμε το μεγάλο ε, ε διοικητικό άχθος. Ε, θα πρέπει να δούμε τι είδους, για τι προγράμματα μιλάμε στην πραγματικότητα, αλλά δίχως άλλο Είμαστε ανοιχτοί στο να εξεταστούν αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την γνωμοδότηση αυτή που υποστηρίζει την πρόταση αυτή που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, το να δείξουμε ένα ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά και χαίρομαι που η Επιτροπή Μεταφορών υπέβαλε μία σειρά από προτάσεις στα πλαίσια της ε, ε, ενιαίας αγοράς και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον έγινε γιατί ένα κοινό ε, και ένα κοινό σχέδιο με την Επιτροπή Μεταφορών. Κύριε Κοφεράτη, πολύ σύντομα μία ανακεφαλαίωση. Νομίζω ότι θα γίνουν σεβαστές οι επιθυμίες και οι ανάγκες των συντονιστών. Θα ήθελα τώρα ε, για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα θετική στάση σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της συζήτησης. Μερικές φορές τα θέματα ουσίας θα μπορούσαν να μας χωρίσουν, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Επιτροπή αυτή να υπάρχει πάντοτε αυτό το κλίμα. Κλίμα που καταγράψαμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο σε διαφορά τις σχέσεις και με την Επιτροπή. Ήμουν δήμαρχος μιας πόλης και ξέρω ότι η κατασκευή ενός δρόμου ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντί για το τραμ, αντί για το σιδηρόδρομο, αντί για τον αυτοκινητόδρομο, ε, ε, όταν έχουμε να κάνουμε με τρένο, με αυτοκινητόδρομο κτλ. οι δυσκολίες αυξάνονται. Προσπάθησα λοιπόν να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της επίλυσης των προβλημάτων που πραγματικά ε, ταλαιπώρησαν ε, πάρα πολλές ε, φορές ε, είναι θέματα που εμφανίζονται και καλούμε θα τα επιλύσουμε. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των συντονιστών και η εκ των προτέρων συζήτηση με τη στην τοπική κοινωνία. Αν είχαμε μπροστά μας ένα πράσινο λιμόνα τα πάντα θα ήταν εύκολα. Αλλά ε, το να κατασκευάσει κανείς ένα δρόμο εκεί που ζουν άνθρωποι και που είναι υποχρεωμένοι να παραιτηθούν από τις καθημερινές τους ε, ε, συνήθες είναι ένα εγχείρημα που πολύ συχνά έχει και ένα πολιτικό κόστος όταν ε, κινηθεί κάπως άνετα. Αυτό ε, το λέω στους συναδέλφους και θα πρέπει να σας πω ότι έχω μια ιδιαίτερη αιμονή για αυτά τα θέματα από τη στιγμή που έχω μια κάποια εμπειρία σε αυτό το τομέα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με τις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Πιστεύω... Α, ε, ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι... Μισό λεπτό να ελέγξω. Ναι, προθεσμία είναι τον Ιούλιο για την υποβολή των τροπολογιών. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε όσο χρόνο φτάνει για να μπορέσουμε να ε, δουλέψουμε χωρίς να αγχωθούμε. Ναι, ναι η 10η Ιουλίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, 10 ιουλιου ειναι η προθεσμια καταθεση τροπολογιων 10 ιουλιου το μεσημέρι. Θα έχουμε επί τα δύο δυνατότητες να συζητήσουμε τις τροπολογίες πρώτα στις 6 Σεπτεμβρίου και τις συμβαστικές τροπολογίες 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Επομένω θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή δουλειά στο τέλο, την οποία θα παρακολουθήσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έγκριση θα γίνει στι 10 ή 11 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μα και αυτό μα επιτρέπει να έχουμε πολύ χρόνο σε σχέση με την Επιτροπή Μεταφορών, η οποία θα εγκρίνει την έκθεση στι 5 Νοεμβρίου. Κύριε Κοφεράτη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται το δημόσιο τμήμα τη συνεδρίασή μα στο σημείο αυτό και θα ξεκινήσουμε στι 5 η ώρα τώρα, δηλαδή την συνεδρία των συντονιστών. Θα σας δω, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 9 το πρωί, αύριο, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη θα είναι η δική μου έκθεση για τα σκάφη ψυχή και ατομικά σκάφη. Ελπίζω λοιπόν να είστε εδώ, θα είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Θα μιλήσουμε για κάποιε νέε κατηγορίε σκαφών και νέα σχέδια σκαφών. Αν θέλετε λοιπόν εξασφαλίσετε την αυτική ασφάλεια κατά τη διάρκεια των διακοπών σα να είστε εδώ πέρα αύριο σε 9 ώρα το πρωί. Και στι 9.30 αύριο θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ πολύ. Λύεται συνεδρίαση.